Οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων μπορούν να θέτουν ερωτήσεις για ένα λεπτό και να παίρνουν απαντήσεις αντίστοιχες χρονικά. Κάθε πρόεδρος της πολιτικής ομάδας, εφόσον το θεωρεί κατάλληλο, μπορεί να θέσει μια συμπληρωματική ερώτηση, η οποία και αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα και πρέπει να έρθει και μια σύντομη επίσης απάντηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίσεως αυτής της συνεδρίασης θα υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα. Τα θέματα είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στις ερωτήσεις οι οποίες είναι καταγεγραμμένες. Η πρώτη ερώτηση προέρχεται από τον κύριο Ζωζεφ Ντόλ. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε Μπαρόσο, η πολιτική μου ημάδα και οι περισσότεροι από εμά εδώ έδωσαν τεράστιους αγώνες για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και είναι πλέον σε ισχύ εδώ και τρει μήνε. Αυτό έγινε για να έχει στη διάθεσή τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μια άξια πολιτική της επίπεδο προσδοκιών. Ακολουθούμε τον σωστό δρόμο, τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μπορούν να ακουστούν, το ζητούν αυτό. Η φωνή τους πρέπει να ακουστεί. Η Ευρώπη θα πρέπει στην παγκόσμια σκηνή να δείξει ποιες είναι οι αξίες της και ποια είναι η φωνή της. Και τι γίνεται με την εξωτερική υπηρεσία την οποία θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα πρέπει επίσης ε, να είμαστε συνδεδεμένοι με τη διαδικασία διαμόρφωσής της. Έτσι κι αλλιώς, όντας η ούσα μάλλον υπεύθυνη αρχή επί του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται και νομικά στη διαδικασία αυτή. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να είναι πλήρως υπεύθυνη και υπόλογη και πολιτικά και οικονομικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε Ντόλ. Απαντά ο Πρόεδρος Μπαρόσο. Ξέρετε ότι η δημιουργία της εξωτερικής κοινή υπηρεσίας είναι μια βασική ρήτρα της νέας συνθήκης και θα ε, συνδράμει την ύπατη εκπρόσωπο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Θα επιτρέπει στα διάφορα κράτη-μέλη να συντονίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμφωνήσει φυσικά με τη συμφωνία του Συμβουλίου για τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας. Θα υπάρξει μια ειδική συνεδρίαση του συνόλου των επιτρόπων την επόμενη Πέμπτη. Είμαι υπέρ μια ισχυρή ευρωπαϊκής Υπηρεσία, η οποία θα λειτουργεί συντονιστικά και θα συνδέει με χρήσιμο τρόπο τα διάφορα κράτη-μέλη με τις κεντρικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σώμα αυτό θα βρει την σωστή του θέση στα πλαίσια της κοινοτικής αρχιτεκτονικής υπό την καθοδήγηση της υπάτου εκπροσώπου η οποία ως ούσα και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνη για τα θέματα της εξωτερικής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ο κύριος Σούλτς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο, η κρίση του ευρώ ξεκίνησε από μη ορθά στοιχεία που έδινε η Ελλάδα. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν εσείς, μπορείτε να επιβεβαιώσετε κύριε Μπαρόζο, ότι ποτέ σε καμιά στιγμή προτού η ελληνική κυβέρνηση υποβάλει τα νεότερα στοιχεία για το έλλειμμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα σε εσά, εσείς, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής σας Επιτροπής για τα πραγματικά στοιχεία είχατε ήδη ενημερωθεί. Δεύτερον, Μπορείτε να επαληθεύσετε, να επιβεβαιώσετε ότι γενικό ε, διευθυντή τη Ευρωστάτ, ο κύριος Ράντεμαχερ, ήδη το 2004 και ήδη το 2005 είχε εκφράσει σημαντικές αμφιβολίες για τα στοιχεία που υπέβαλε η Αθήνα. Και τι κάνατε εσείς τότε, ώστε η Ευρωστάτ να υποστηριχθεί κατά την συλλογή στοιχείων. Τρίτον, αληθεύει ότι οι επιθεωρητές της Ευρωστάτ σας ενημέρωσαν ότι υπήρχαν σημαντικές αμφιβολίες για τα στοιχεία που υπέβαλε η Αθήνα. Ε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς επειδή υπήρχαν αμφιβολίες όσον αφορά τα ελληνικά στοιχεία από πλευρά τη Επιτροπή ο κ. Αλμούνια που ήταν αρμόδιο για αυτό το χαρτοφυλάκιο τα τελευταία χρόνια με μεγάλη αμεροληψία και αντικειμενικότητα και σε βάθο γνώση Γι' αυτό όχι μόνο αναφερθήκαμε σε αυτό το σημείο επανειλημμένα έναντι των ελληνικών αρχών, αλλά υποβάλαμε και ένα κανονισμό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως πρόταση, προτείνοντας να δοθούν στην Ευρωστάτ ελεγκτικές εξουσίες. Δυστυχώς αυτή η πρότασή μας απορρίφθηκε από τα κράτη-μέλη. Δεν επιθυμούσαν τα κράτη-μέλη να λάβει η Ευρωστάτ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες εξουσίες, περισσότερες αρμοδιότητες, ώστε να εμβαθύνουν τους ε, εθνικούς λογαριασμούς της Ελλάδας. Και πρέπει να σας πω ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να υποβληθεί και πάλι εκ νέου αυτός ο κανονισμός ως πρόταση. Και η πληροφορία μου είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις χώρες που είχαν καταψηφίσει θεωρούν ότι αυτή τη φορά είναι πιο έτοιμες και θα ψηφίσουν υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας. Panie Przewodniczący, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów. Eksonomatos tis ομάδας των Φιλελευθέρων Δημοκρατών. Vielen Dank, Ευχαριστώ πολύ. Το κατανόησα. Ο κύριος Αλμούνια λέει ήταν ο αρμόδιος. Εγώ ζήτησα για τη δική σας τοποθέτηση, αλλά θα μου πείτε αμέσως βέβαια τι κάνατε ο ίδιος. Σας κατάλαβα καλά κύριε Μπαρόζο ότι η ευθύνη για την ελληνική κρίση βρίσκεται στα κράτη-μέλη. Λέει, διότι αυτά λέει αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις προτάσεις σας. Και παρακαλώ να μας πείτε ποιοι αρχηγοί κυβερνήσεων, ποια κράτη-μέλη ήταν αυτά που ήταν εναντίον. Ευχαριστώ. First of if you ask me about the αν θέλετε να μου πείτε ποιος φταίει, εγώ δεν, ε, ε, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πέρα από το ότι οι ελληνικές αρχές δεν σεβάστηκαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος κ. Σαλμούνια με την πλήρη υποστήριξή μου και το συνόλου του Επιτρόπων έκανε τη δουλειά του με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο. Και το θέμα αυτό είχε συζητηθεί επανειλημμένα Θυμίζω ότι πολλά κράτη-μέλη είχαν ε, καταψηφίσει την πρόταση που είχαν κάνει, δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά η Γερμανία σαν παράδειγμα το είχε καταψηφίσει. Και οι Γερμανοί αυτή τη φορά μου είπαν ότι θα υπερψηφίσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα υπάρχει μια συνένεση σύμφωνα με την οποία απαιτείται μια ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έγιναν κάποιες προτάσεις και από την γερμανική πλευρά σχετικά με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Έγιναν και κάποιες άλλες προτάσεις και επιλογές για την δημιουργία μιας υπηρεσίας διαχείρισης χρέους η δημιουργία των ευρωομολόγων ή και η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας αξιολόγησης ή βαθμολόγησης. Τα πράγματα λοιπόν φαίνεται ότι κινούνται και κινούνται σχετικά γρήγορα σε αυτή τη φάση. Τρεις λοιπόν πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί μια συγκεκριμένη προτάσεως για τη δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Δεύτερον, είναι αλήθεια όπως είπε η κυρία Μέρκελ, αν και εγώ αμφιβάλλω, ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει συνθήκη για να γίνει κάτι τέτοιο. Για να γίνει δηλαδή το τομείο αυτό. Και τρίτον, συμφωνείτε ότι το ταμείο αυτό δεν είναι παρά ένα πρώτο βήμα για να υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα έχουμε όλοι ανάγκη. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, η ιδέα προτάθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών μάλλον της Γερμανίας. Χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Όμως συμβάλλει στη σημερινή συζήτηση γύρω από το ευρώ και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο είναι μια μακρόπνοη πρόταση που ενδεχομένως χρειάζεται μεταβολή της συνθήκης. Αυτό το οποίο επεξεργαζόμαστε είναι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ε, παρακολούθησης των κρατών. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ακριβώς το σχήμα. Γενικά, όπως είπατε, υποστηρίζουμε τα πάντα που ενισχύουν την οικονομική δημοσιονομική διακυβέρνηση. Αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες και να υποβληθεί πρώτα στην κατάλληλη στιγμή. Τούτου λεχθέντος, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο δεν θα επέλυε το επίγον πρόβλημα της Ελλάδος. Είναι ξεχωριστό ζήτημα που πρέπει να αναλυθεί περισσότερο και είναι πιο μακρόπνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο της Κομισιόν για την απάντηση που μου έδωσε. Συμφωνώ μαζί του το Ταμείο Περσέ δεν μπορεί να επιλύσει άμεσα προβλήματα. Ε, η ερώτησή μου είναι η εξής, μάλλον η πρόταση μου είναι η εξής εξετάζοντας το θέμα η Κομισιό να εξετάσει και τις διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Το νομισματικό ταμείο, τα ευρωομόλογα που είναι μια άλλη ιδέα που μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα είναι ο οίκος αξιολόγησης, ε, η υπηρεσία αξιολόγησης που προτείνει ο πρόεδρος του Eurogroup ώστε να μην εξαρτώμαστε από τους ξένους οίκους αξιολόγησης και υπάρχει Υπάρχουν και άλλες ιδέες. Η σκέψη μου λοιπόν είναι όλες αυτές, ε, να γίνει μια σύνθεση αυτών των ιδεών και να έρθει η Κομισιόν με μια συνεκτική πρόταση. Μα ακριβώ λέει ο πρόεδρος για να αποφύγουμε αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα ε, κάνουμε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν προτάσεις διαφορετικές από την ίδια κυβέρνηση καμιά φορά. Γι' αυτό δεν θέλουμε να επισπεύσουμε, δεν θέλουμε να βιαστούμε ο Επίτροπος, ο Λιρέν, το είπε ήδη δημόσια. Ετοιμάζουμε μία ανακοίνωση για τον συντονισμό της ενισχυμένης οικονομικής πολιτικής και την παρακολούθηση, την επιτήρηση κρατών μέσα στο πλαίσιο του ευρώ και ακόμη και ευρύτερα μέσα στο πλαίσιο ίσως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επεξεργαζόμαστε αυτή την ανακοίνωση και δεν πρέπει κάθε μέρα να ανακοινώνουμε και μια νέα πρόταση. Εργαζόμαστε με αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρεμπέκα Χάρμς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεδομένης της κατάστασης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πραγματική αγορά ή ανάγκη για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων πατατών και υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει. Σα ερωτώ, γιατί με τόση μεγάλη βιασύνη και πίεση μεριμνήσατε η γενετικά τροποποιημένη πατάτα με γοργέ συνοπτικέ διαδικασίε να εγκριθεί μια και δεν υπάρχει και ανάγκη η ζήτηση. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε σε σχέση με τον νέο Επίτροπο για θέματα υγείας. Πώς τον καταφέρατε τις επιφυλάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας για τις δοκιμές να τις αγνοήσει. Γιατί δεν αναμείνατε μέχρι ότου να υποβληθεί η νέα πρόταση, η νέα οδηγία που εκπονείται, βρίσκεται υπό εκπόνηση αυτή τη στιγμή για την αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά την βιοπικιλότητα και τη βιόσφαιρα γενικά για, από πλευρά των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και φυτών. Και το όριο μόλυνσης ή ε, επιμόλυνσης ε, τροφίμων ε, που μέσω αυτών των διαδικασιών έχει αυξηθεί σε 0,9% είναι μια στρατηγική αντιμετώπιση κινδύνου που δεν είναι είναι αποδεκτή από τους πολίτες μας καθόλου. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Είδαμε την διαμαρτυρία σας. Λήφθη υπόψη. Well, Mr. President, please, yours. Uh, Η Κομισιόν αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει δίνοντας άδεια σε αυτό τον γενετικά τροποποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουμε. Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να σεβόμεθα και να λέμε ναι ή όχι. Ε, υπευλήθη μία προσφυγή και η ΕΦΣΑ, ο εξάρτητος οργανισμός ασφάλειας τροφίμων, εξετάζει την υπόθεση. Θέλουμε να βεβαιωθούμε για την αξιολόγηση παρουσίας ανθεκτικού στα αντιβιωτικά οργανισμού. Μετά την εξέταση δεν υπήρξαν επιστημονικοί λόγοι σύμφωνα με την ανεξάρτητη υπηρεσία για ανατροπή. Συνεπώς έχουν εξεταστεί όλα τα επιστημονικά θέματα και ουσιαστικά περίμενα συγχαρητήρια από σας διαμαρτυρίες από το ακροατήριο, διότι έχω ανακοινώσει ότι η Κομισιόν έχει την πρόθεση να προτείνει να δώσει στα κράτη-μέλη την δυνατότητα, αν θέλουν, να καλλιεργήσουν τις, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό είναι η λογική θέση όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Ορισμένα κράτη ευνοούν και ορισμένα κατακρίνουν. Η κυρία, η κυρία περώσει. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μου δώσατε καμία απάντηση στο ερώτημα για την ανάγκη ζήτηση για αυτή τη γενετικά τροποποιημένη πατάτα που μόνο άμυλο θα προσφέρει, θα δίνει. Υπάρχουν εναλλακτικέ άλλες δυνατότητες. Γιατί να υπομισθούμε τέτοιο κίνδυνο. Και δεύτερον, το επίπεδο ρήπανσης ή μόλυνσης 0,9%. Ε, έχουμε συζητήσει για τις ε, ε, τιμές αυτές και ακριβώς για τις ε, ζωοτροφές και για τα τρόφιμα αλλά και για τα αντιβιωτικά. Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα σε σχέση με την παρόντα. Δεν είπατε τίποτα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Θέλω να μου πείτε, θα υπάρξουν περαιτέρω εγκρίσει χωρί την οδηγία τη ΕΦΣΑ και χωρί σύσταση από πλευρά αυτού του οργανισμού, αν θα πρέπει να δοθούν άδειε όσον αφορά τον αραβόσιτο, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Not Well, Mr. President, uh, seeing, uh, Χαίρομαι για τον ενθουσιασμό της πολιτικής σας ομάδας, σας συγχαίρω για τις εκδηλώσεις αυτές, έχετε σαφέστατες θέσεις κατά. Κατά οποιασδήποτε μορφής γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Εγώ δεν έχω καμία θέση υπέρ ή κατά σε αυτό το θέμα. Εξαρτάται από τις γνωμοδοτήσεις οι οποίες μου δίδονται από τους εμπειρογνώμονες της ΕΦΣΑ. Δεν έχω καμία προκατάληψη υπέρ, καμία προκατάληψη κατά των γενετικά τροποποιημένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη συγκεκριμένη θέση να ακολουθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων. Δεν συζητάμε τα θέματα τα γενετικά τροποποιημένα σε ιδεολογικό επίπεδο. Λαμβάνουμε τις θέσεις μας επί τη βάση των ανεξαρτήτων θέσεων των εμπειρογνωμόνων. Όχι γιατί τα γενετικά τροποποιημένα είναι, είναι απαραίτητα αλλά γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποδείξεις που να δείχνουν ότι είναι επικίνδυνες για την υγεία ή για το περιβάλλον. Λοιπόν, και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που έχουμε, στα πλαίσια του ΠΟΕ, εγκρίνουμε τα προϊόντα αυτά εφόσον δεν υπάρχει τίποτα επιστημονικά το οποίο να μας το απαγορεύει. Διακόπτεται ο πρόεδρος της Επιτροπής από τον πρόεδρο Μπούζεκ για την ομάδα των μεταρρυθμιστών και συνταρρυθμιστών μεταρρυθμιστών Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ε, υπόσχομαι ότι σε σχέση μετά από τα γενετικά τροποποιημένα θα θίξω ένα πιο απλό θέμα, λιγότερο περίπλοκο εννοώ. Όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, κάνουμε λόγο και αυτό είναι σωστό και θεμητό για την σημερινή οικονομική, χρηματοοικονομική κρίση. Και είμαι έχω τη βεβαιότητα ότι τα κράτη-μέλη ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν όσον αφορά την απασχόληση για τους πολίτες τους από ότι για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τις γενετικά τροποποιημένες πατάτες. Αφενός από τη μια πλευρά η Ευρωβουλή τοποθετείται πάντα υπέρ μιας ισχυρής διακυβέρνησης και ανάληψης δράσης γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά λέω, λέμε εμείς οι συντηρητικοί ότι δεν είναι τέτοια μέτρα που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης αλλά τα μέτρα από πλευρά επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσει απασχόληση, οι ίδιε οι επιχειρήσει. Έχω τι εξή ερωτήσει προ εμά. Ποια είναι η ανεξαρτησία που αφήνεται σε σχέση με τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσκολίες. Δεύτερον, μπορείτε να υποσχεθείτε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία θα μειωθεί διότι επιβαρύνει, είναι βάρος για την οικονομική ανάπτυξη. Μπορείτε να συμφωνήσετε μαζί μου ότι λιγότεροι κεντρικοί κανόνες και λιγότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι η καλύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σεβόμαστε απολύτω την ποικιλομορφία των κρατών μελών. Γι' αυτό στη στρατηγική του 2020 αποσαφηνίζουμε τα πράγματα και δημιουργούμε μηχανισμούς όπως η πολιτική, η κοινωνική πολιτική. Δεν είναι όλες οι πολιτικές οι ίδιες, το είπαμε αυτό. Θέλουμε όμως ισχυρότερη διακυβέρνηση διότι αν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν κάποιες πολιτικές δεν θα έχουν την, τον ίδια δύναμη να συζητήσουν ε, επίσης βάσεως με μεγάλους ε, μεγάλες χώρες όπως η ΙΠΑ και η Κίνα, μόνοι τους πάντα. Όσον αφορά το θέμα της μείωσης του αρχικού φορτίου, πιστεύουμε σε αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε προοδευτικά και να αποφεύγουμε νομοθετήματα όταν αυτά δεν είναι απαραίτητα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Λότερο Μπίσκι, παρακαλώ, Ηνωμένη Αριστερά. Κύριε Μπαρόζο, την προηγούμενη εβδομάδα εσείς υποβάλλατε την πρότασή σας για μια οικονομική στρατηγική. Αχρειάζονται όμως και λείπουν από την ε, σημαντικές στοχοθετήσεις. Το Συμβούλιο επέβαλε στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα λιτότητας που αυτούς τους στόχους τους θέτουν στο επίπεδο του ανέφικτου πλέον. Και σε σχέση με το ΑΕΠ που θα πρέπει να ε, είναι στο, το έλλειμμα στο 3% όμως σε σχέση με το αποτυχημένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης ενώ ταυτόχρονα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν, θέτουν το αίτημα για ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο ή Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, η οικονομική διακυβέρνηση θα επανεξεταστείτε και θα επανεκπονήσετε τους στόχους 2020 ώστε να ενταχθεί η ιδέα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης και να αποφευθεί το ντάμπινγκ, το φορολογικό και να μπορέσουν στρατηγικές ευρωπαϊκές να ξεκινήσουν. Άμεσα με τα κράτη-μέλη από κοινού θα λάβετε μέτρα ώστε η κερδοσκοπία των τραπεζών κατά του ευρώ να σταματήσει επιτέλους που σώθηκαν αυτές οι τράπεζες με χρήματα φορολογουμένων πρόσφατα εξάλλου. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τη θέση της Ελλάδας, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσει το έλλειμμα φέτος. Είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα δομικά προβλήματα, τα διορθωτικά. Ταυτόχρονα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα της ζώνης ευρώ. Συνεργάζεται η Κομισιό με τα κράτη-μέλη για να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που η Ελλάδα θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί. Και θα είναι σύμφωνος ο μηχανισμός με τις συνθήκες και θα είναι αυστηροί οι κανόνες. Θα έχουμε ένα πλαίσιο για συντονισμένη βοήθεια και την υποστήριξη βεβαίως των κρατών της Ευρωζώνης. Αυτά μπορώ να σας πω για την Ελλάδα και για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Όσον αφορά τις προτάσεις του Unicredit δεν πρέπει να μεταβληθούν. Πρόκειται να συζητηθούν οι προτάσεις από το Συμβούλιο και από το Ευρωκοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι αυτή η συζήτηση θα αποβεί καρποφόρα. Κύριε Πρόεδρε, δεν με ικανοποιεί απόλυτα αυτή η τοποθέτηση. Το θέμα, το ερώτημα είναι το εξή. Το ότι με χρήματα φορολογουμένων έγιναν πράξεις κατά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου και υπάρχει κερδοσκοπία με αυτά τα κονδύλια. Τα χρήματα των φορολογουμένων προέρχονται και από... Ε, γι' αυτό, γι αυτό το σκοπό δεν διατέθηκαν και δεν γίνεται τίποτα. Είμαι απογοητευμένος ότι τόσα λίγα έχουν γίνει και γίνονται ώστε συγκεκριμένα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάψουν ή να σταματήσουν επιτέλους ώστε να πάψει αυτή η κερδοσκοπία και να επικεντρωθούμε στην προσπάθεια της ανάκαμψης. Ευχαριστώ. Oh, uh, Σε σχέση με την κερδοσκοπία, είμαστε σαφείς ότι τα τρέχοντα προβλήματα στην Ελλάδα δεν προέκυψαν από την κερδοσκοπία. Βασικά προήλθαν από υπερβολικές δαπάνες και μη τήρηση του πλαισίου σταθερότητας, ε, υπερβολικό χρέος δηλαδή, υπερχρέωση. Βεβαίως στη συνέχεια οι κερδοσκόποι πράγματι ε, δημιούργησαν προβλήματα για το δημόσιο χρέος. Χρειάζονται βεβαίως τροποποιήσεις και μεταβολές στην αγορά, χρειάζονται δράσεις από την Κομισιόν το 2009. Ξεκίνησε η Κομισιόν ένα πρόγραμμα για, να γίνει η αγορά των derivatives των παραγόγων ε, σταθερή. Προχώρησε με μια οδηγία. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα υποβάλει αυτή την ε, οδηγία για την, ε, τον έλεγχο των κινδύνων. Χρειάζεται επίσης να ασχοληθούμε με τα swaps σε σχέση με τα κρατικά χρέη και δεν είναι αιτιολογημένο να, ανεβαίνουν η να ανεβαίνει η ασφάλιση κινδύνου αλλά βράχει πρόθεσμα πρέπει να πετύχουμε συντονισμένο τρόπο ενέργειας των κρατών μελών και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν θα εξετάσει προσεκτικά το ενδεχόμενο απαγόρευσης α, της διαπραγμάτευσης των swaps για τα κρατικά χρέη. Βεβαίως είναι να οι αγορές. Θα φέρουμε αυτό το θέμα στην ομάδα των 20 και θα το θέσουμε και στις διμερείς μας επαφές, ειδικότερα με τσίπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν σας διέκοψα γιατί ήταν πολύ σημαντική απάντηση. Ε, η απάντησή σας πήρε κάπως περισσότερο χρόνο από αυτόν ο οποίος προβλέπεται η κυρία Νίκη Τζαβέλα. Ερώτηση την οποία θα έθετα. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ω Ελληνίδα Ευρωβουλευτής επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Η δοκιμασία αυτή την οποία περνάμε αυτή την περίοδο και για την οποία είμαστε υπόλογοι είναι ένα πολύ καλό τεστ αντοχής και πειθαρχία για την Ελλάδα κύριε πρόεδρε χάρηκα πάρα πολύ που αναφέρατε τους g twenty σαν μια ομάδα στην οποία θα φέρετε το θέμα των swaps. η ελλάδα πέρα των δικών της σφαλμάτων χτυπήθηκε σκληρά από την κερδοσκοπία των αγορών. προτίθεστε πραγματικά και θα ήθελα κάπως να το αναπτύξετε αυτό στο πλαίσιο των g 20 να ηγηθείτε πρωτοβουλίας για τη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων όσον αφορά τις ανοιχτές ακάλυπτες πωλήσει και τα credit default swaps. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα προηγουμένως, το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας προέρχεται από το υπερβολικό χρέος της χώρας αυτής. Προφανώς και έχουν υπάρξει και κερδοσκοπικέ επιθέσεις, ακριβώς όμως επειδή είδαν ότι υπήρχαν οι δυνατότητες. Προφανώς και πρέπει να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Έχει ανακοινώσει εξαιρετικά σημαντικά μέτρα η ελληνική κυβέρνηση και τα υποστηρίζουμε. Σχετικά με το ευρύτερο θέμα είπα ότι θα εξετάσουμε εκ νέου το θέμα της απαγόρευσης κερδοσκοπικών συναλλαγών γύρω από τα CDS σε σχέση με το δημόσιο χρέος χωρών. Το θέμα της διαφάνειας ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές και γύρω από το θέμα της πρόσβασης σε πληροφορίες για τέτοιου είδους πρακτικές θα τεθεί και στην ομάδα των 20 και σε άλλα φόρα. Και επαναλαμβάνω, ότι οργανώνεται μία συνάντηση από τον Επίτροπο Μπαρνιέ με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτές τις επιθέσεις των κερδοσκόπων, ε, επιθέσεις στα χρέη των χωρών. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα swaps και πώς λειτουργούν οι αγορές των CDS και να δούμε αν υπάρχουν θέματα αμφισβητούμενων πρακτικών. Ο κύριος Μπαρνιέ θα το εξετάσει και αυτό. Ε, Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε αυτό που λέτε για τον μηχανισμό καταπολέμησης της κερδοσκοπίας. Αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για να ξέρω όταν θα βγούμε για δανεισμό στη διεθνή αγορά αν θα έχουμε κάποια στήριξη από αυτό το μηχανισμό. Το είπα και θα το επαναλάβω. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα παρουσιάσει τις προτάσεις του πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα κάνει κάποιες προτάσεις για αλλαγές σχετικές με την οδηγία για τα παράγωγα και σε σχέση με την οδηγία για τις καταχρήσεις. Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις αυτές θα βελτιώσουν τη διαφάνεια των αγορών και θα μειώσουν τους κινδύνους. Το θέμα των CDS θα τεθεί στη συνάντηση του G20 τον μήνα Ιούνιο. Σας ευχαριστούμε κύριος Ντάνιελ Βαντερστερ παρακαλώ. Στο πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο, ανοιχτό πλαίσιο και διαφάνεια, αρχές κάθε δημοκρατίας που σέβεται τον εαυτό της. Όταν οι κυβερνώντες στις δαπάνες τους δεν ελέγχονται από τους πολίτες, τότε μπορεί να υπάρξει μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα διαφθοράς και πλουτισμού. Αυτό το είδαμε και πέρσι στην Μεγάλη Βρετανία. Στον Ολλανδικό τύπο είδαμε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2009 είχε 730.000 λέει ευρώ δαπάνες ε, ταξιδίων και ε, αποστολών. Είναι τεράστιο αυτό το ποσό, έτσι δεν είναι. θα πόσα θα έπρεπε να δίνετε κάθε μέρα, μερικές χιλιάδες ευρώ για να φτάσετε σε αυτό το ποσό. Τώρα, χωρίς αστεία, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχει εσωτερικός έλεγχος και κάποιοι ελεγκτέ ε, που όλα αυτά ε, τα έχουν επιβεβαιώσει. Ζητώ από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έναντι του κ. Μπαρόζο αυτό το, αυτή η πρακτική να σταματήσει πια να υφίσταται και όλε οι δαπάνε να είναι ανοιχτέ και να μπορούν να ελεγχθούν δημόσια. Ευχαριστώ. The... Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή. Έχετε το. In fact, um, the so expenses are expenses... Οι δαπάνες αυτές είναι δαπάνες που αφορούν γενικά τις υπηρεσίες τη Επιτροπής, τα ταξίδια των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα δικά μου και των άλλων επιτρόπων. Αν συγκρίνετε τα ποσά αυτά με αυτά τα οποία δαπανούν πολλές φορές κυβερνήσει, ή ηγεσίε κυβερνήσεων κτλ. θα δείτε ότι τα ποσά αυτά είναι πάρα πολύ λίγα, πάρα πολύ μικρά. Ο προπολογισμό για το σύνολο των επιτρόπων καθορίζεται από τις αρμόδιες δημοσιονομικές αρχές, είστε τμήμα αυτής της αρχής και υπάρχουν προσαρμογές ανά πενταετία μόνο σε σχέση με τον πληθωρισμό. Πιστεύουμε ότι είναι έλογες οι δαπάνες αυτές και είναι ανάλογες με τη σημασία των θεμάτων τα οποία επιδιώκουμε. Προφανώς και χρησιμοποιούμε την πλήρη διαφάνεια. Είναι γνωστά τα στοιχεία μας και προς το ελεγκτικό συνέδριο και προς τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου. Σας ευχαριστούμε. Και πάλι λοιπόν. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπαρόζο, λέτε, η Ευρωβουλή λέει αυτές τις δαπάνες μπορεί να τις δει. Είναι όμως ανοησίες αυτές όλα γίνονται εγκρυπτό και παραβίστο. Όλα γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο, θα έλεγε κανείς, μυστικότητας. Θα πρέπει αυτά, αν τα λέτε σοβαρά, να γινόντουσαν δημόσια, διότι διαφορετικά ομολογείται ότι γίνονται εγκρυπτό και παραβίστο. Δεν κατανοώ αν αληθεύουν αυτά τα οποία λέτε, γιατί αυτά τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται. Φοβόσαστε την οργή και την αντίδραση των πολιτών. Σε ένα σύστημα που διέπεται από τον νόμο τηρούμε τους κανόνες, σεβόμαστε τους κανόνες. Γίνεται φασαρία στο ακροατήριο χωρίς κάποιον συγκεκριμένο μιλητή. Ο πρόεδρος Μπαρόζο θα απαντήσει, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σε ένα δικαϊκό σύστημα κανείς τηρεί τους νόμους και τις διατάξεις. Την ανάλυση προθέσεων ε, να γίνεται ανάλυση προθέσεων είναι άδικο. Δεν μπορείτε να αποδώσετε καμία πρόθεση σε μένα ή στην Κομισιόν όσον αφορά την τήρηση του δικαίου. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ των υποχρεώσεων ε, τήρησης του δικαίου και των δημαγωγικών επιθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και γενικά όλα τα θεσμικά όργανα είναι πάρα πολύ διαφανή. Δεν δέχομαι λοιπόν τη δημαγωγική σας λαϊκίστικη κριτική. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Ολοκληρώσαμε έτσι τον πρώτο γύρο ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γενικής φύσεως ερωτήσεις. Και τώρα θα επικεντρωθούμε σε ένα ειδικό εξειδικευμένο θέμα που είναι η εφαρμογή της νέας συνθήκης. Και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο πρώτος ομιλητής θα είναι ο κύριος Μέσσον. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι δεν θα παρεκκλίνω από τα ερωτήματα τα οποία πρέπει τώρα στη συνέχεια σε αυτό το γύρο να διατυπωθούν. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Μπαρόζο και εμείς και εγώ συμφωνούμε για το ότι η διαπίστωση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί και αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει στην Ερυθρέα. Και από το 2009 έως το 2013 προβλέπεται ένα μεγάλο ποσό 100 ευρώ αναφέρεται. Θα έλπιζα ότι γνωρίζει ο κύριος Μπαρόζο πού θα δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως όμως θα έπρεπε να τοποθετηθεί και να γνωρίζει τα σχετικά ο κύριος Μπαρόζο για την Ερυθρέα. Διότι συχνά η Ερυθρέα δεν αναφέρεται όταν κάνουμε λόγο για ολοκληρωτικά καθεστώτα. Άλλες χώρες αναφέρονται και όχι η Ερυθρέα. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω την άποψη του κυρίου Μπαρόζο για την Ερυθρέα. Ευχαριστώ. Thank you for recognizing that the Commission Ευχαριστώ ότι αναγνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτό αυτή και στι εξωτερικέ μα σχέσει. Δεν είναι δυνατόν να ε, αποφύγουμε να γίνεται αυτό. Και υπάρχουν δυστυχώ χώρε ε, που δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. παρόλα αυτά πρέπει να καλλιεργούμε τη σχέση μα με τι χώρε αυτέ. Η περίπτωση τη Ερυθρέα είναι μια τέτοια περίπτωση όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία υφίσταται εκεί και μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνα με κάποιους ε, σχολιαστές ε, ως ε, μια καταραίουσα χώρα επειδή υπάρχει διαδεδομένη βία, δεν υπάρχει καθεστώς ένομης τάξης και πάρα πολύ Πάρα πολλές φορές ούτε καν οι, αρχές, οι κρατικές αρχές δεν μπορούν να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όμως την κατάσταση σε όλες τις χώρες που μπορούν να θέσουν ενδεχόμενα ένα πρόβλημα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. Παν Άρτουρ Ζασάντα, ένα μινούτα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αρτούρ Ζασάντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Μέσα στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο θέμα των σαρωτών σώματο στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια Μία από τις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν πρέπει λοιπόν να δεχθούμε μια κατάσταση που δημιουργείται μια χήμερα, μια φρούδα ελπίδα ασφάλειας και ελευθερίας, ενώ παραβιάζονται δικαιώματα της ιδιωτικής σφαίρας και ζωής. Η κατάσταση σαρατών σώματος είναι παρόμοια με εκείνη που ζήσαμε και βιώσαμε κατά τη διάρκεια της ε, νέας ε, επιδημίας γρήπης που είχε σημειωθεί. Επενδύθηκαν μεγάλα ποσά σε σχέση με εμβόλια τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Και σήμερα το ίδιο φαίνεται να επαναλαμβάνεται ότι ασκείται δηλαδή πίεση για να επιβληθούν να λειτουργήσουν οι σαρωτές σώματος. Θα ήθελα να ακούσω την δική σας άποψη Πρόεδρε. Εγώ είμαι απόλυτα κατά των σαρωτών σώματος. Ευχαριστώ. Θα είμαι υπέρ αν συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Διότι πρέπει να έχουμε μια ομαλοποίηση, τυποποίηση των κανόνων ασφάλειας στα αεροδρόμια μας. Τι συμβαίνει σήμερα. Ορισμένα από τα κράτη-μέλη εισάγουν τους αεροτές στα αεροδρόμια. Άλλα κράτη-μέλη δεν τα τοποθετούν αυτά τα μηχανήματα. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν έχει υποβάλει μια πρόταση για τους σαρωτές που απορρίφθηκε. Αυτό έχει προκαλέσει κάποιες ανησυχίες. Πρέπει να βρούμε όμως μια εναρμονισμένη θέση όσον αφορά την χρήση οποιοδήποτε μηχανήματος για λόγους, ασφα... Ε, ε, για λόγους ασφάλειας στα αεροδρόμια. Δεν μπορούμε να έχουμε διακρίσεις όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας στα αεροδρόμια μας. Σας ευχαριστώ. Ο Παντέρεκ Βόγκεν. Η συνθήκη σέβεται τα δικαιώματα των τοπικών αρχών και των περιφερειών στην Ευρώπη. Είναι σημαντικός παράγοντας αυτός όταν ξεκινάτε τις συζητήσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Όταν θα ξεκινήσετε λοιπόν αυτές τις συζητήσεις για την πέμπτη έκθεση συνοχής, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα συνομιλήσετε και με τις τοπικές αρχές και τις περιφερειακές αρχές σχετικά με την ε, μελλοντική πολιτική συνοχής και με το Ευρωκοινοβούλιο. Πρόεδρο Μπαρόζο. Δεν είναι θέμα θεμελιώδων δικαιωμάτων αυτό βεβαίω, αλλά είναι αυτονόητο ότι θα συζητήσουμε με τι τοπικέ και τι περιφερειακέ αρχές. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για μα να έχουμε εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή. Αναγνωρίζεται από τη συνθήκη της Λισαβόνα σαν ένας από τους στόχους. Στην στρατηγική που, εμφαν... Ε, που σας υπέβαλα προ ε, είναι βέβαιο ότι οι περιφέρειες θα μείνουν, ε, μάλλον η Κομισιόν θα μείνει μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής και θα συνεχιστεί αυτό. Σας ανέφερα ήδη ένα έγγραφό μας και βεβαίως θα πρέπει να συμβουλευτούμε και την Επιτροπή Περιφερειών. Η Κατερίν Στίλερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο Μπαρόζο. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο φέρμα την Σκοτία ήρθε σε επαφή ένας κύριος σε σχέση με ένα θέμα στην Ερυθρέα. Υπάρχει εκεί δίωξη των χριστιανών Κατάφερε λοιπόν ένας άνθρωπος να ξεφύγει στην Ιταλία και μετά στη Σκοτία. Τη φρόντισαν εκεί Σκοτσέζοι. Είναι 16 ετών αυτό το κορίτσι. Αντιμετωπίζει περίπτωση απέλασης και θα θέλαμε να βοηθηθεί ώστε να μπορέσει να μείνει στην οικογένεια που την υιοθέτησε. Θέλουμε τη βοήθεια των όλων έχει την υποστήριξη των ΜΚΟ της περιοχής. Τι θα μπορούσε η Κομισιόν να κάνει για να προστατεύσει τα δικαιώματα αυτού του κοριτσιού. Λυπάμαι, αλλά δεν γνωρίζω αυτή την εξειδικευμένη περίπτωση συγκεκριμένα στην Σκοτία. Είναι μια γενική παρατήρηση που πρέπει να κάνω. Αυτή η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να αναμένει κανείς από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα και αν εργάζεται σχετικά σκληρά να γνωρίζει όλα αυτά είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και όμως φυσικά σε σχέση με την έκφραση της δικής μας ε, ε, αίσθηση. Είμαστε αλληλέγγυοι προ οποιοδήποτε άτομο του οποίου τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται ή παραβιάζονται. Δεν έχω όμω περισσότερα στοιχεία. Ευχαρίστω να αντιδράσω γραπτό επιστολή στο θέμα το οποίο θέσατε. Ευχαριστώ. Αλβάρο, παρακαλώ. Εξ ονόματο τη πολιτική μου ομάδα, στι 5 Μαρτίου ο πρόεδρο τη Ιταλική Δημοκρατία Τζόρτζο Ναπολιτάνο υπέγραψε ένα διάταγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, η προεκλογική εκστρατεία να αλλάζουν οι εκλογικοί κανόνες. Ο ίδιος ο Ναπολιτάνο είπε ότι στην πρόταση νόμου το κείμενο το οποίο του είχε υποβληθεί από πλευρά του Συμβουλίου Υπουργών της Ιταλικής Δημοκρατίας δεν παρουσίαζε συνταγματικά προβλήματα. Στο άρθρο 87 το Σύνταγμα της Ιταλικής Δημοκρατίας λέγει ότι οι αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν ισχύ νόμου. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως να λαμβάνει μέρος στη διαδικασία κατάρτισης των νόμων αυτών και συγγραφής των νομικών ρυθμίσεων. Πρόκειται για μια στρέβλωση του δημοκρατικού συστήματος. Το διάταγμα αυτό άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού και έχει δημιουργήσει συνταγματικά προβλήματα. Διακόπτεται η ομιλήτρια. Διαρωτώ με γιατί το κοινοβούλιο αυτό είναι πάντα διατεθειμένο να καταφέρεται εναντίον χωρών που παραβιάζουν τον νόμο αλλά όχι εναντίον των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραβιάζουν τον νόμο. Ενός λεπτού η ερώτησή σας κυρία μου. Παρακαλώ σεβαστείτε τον κανόνα. Για μια ακόμη φορά απαντάει ο Πρόεδρος μη μου ζητάτε να μπω στα θέματα εσωτερικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ευθύνε σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου είτε από τα κράτη-μέλη είτε από τα ευρωπαϊκά όργανα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει θέμα εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αν κατάλαβα καλά από τη δική σα παρουσίαση πρόκειται για ένα θέμα εσωτερικό πολιτικό τη Ιταλίας μπορεί να έχει μια διάσταση σε επίπεδο πολιτικών δικαιωμάτων ή σε επίπεδο κράτους δικαίου, αλλά παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και τις πολιτικές προσωπικότητες των χωρών μελών. Ουρρίκε Λονάτσεκ παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο, η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι το μέχρι σήμερα μόνο διεθνές έγγραφο το οποίο την αρνητική μεταχείριση την απαγορεύει ακόμα και με βάση σεξουαλικούς προσανατολισμούς και επιλογές. Και έναντι των άλλων υπήρων και χωρών του κόσμου το κατάφερε αυτό η Ευρώπη. Το πρόβλημα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι τρεις χώρες, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία και Τσεχία, τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν την θεωρούν άρρηκτα τμήμα της νομοθεσίας τους. Με ενδιαφέρει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι έχετε εσείς υπόψη να κάνετε ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ομοφιλοφίλων να μπορέσουν για όλους να είναι σεβαστά και να είναι σαφέ ότι η ομοφιλοφοβία και ε, η, αντική η αντιμετώπιση με βάση τις ε, σεξουαλικέ επιλογές δεν μπορεί να γίνεται δεκτή πλέον και ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ελεύθερα ελεύθεροι από φόβο και να μπορούν να διαμορφώνουν τις ερωτικές τους σχέσεις ελεύθερα. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Δύο ερωτήματα υπάρχουν εδώ. Δεν γνωρίζω αν μπορώ σε ένα λεπτό να τα απαντήσω. Πρώτον, όσον αφορά αρνητική μεταχείριση σε σχέση με τις σεξουαλικές επιλογέ. Γνωρίζετε ότι η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει μια οδηγία κατά οποιασδήποτε αρνητική μεταχείριση ακόμα και με βάση σεξουαλικές επιλογές και όσον αφορά την απασχόληση. Είμαστε δεσμευμένοι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η υλοποίηση από τα κράτη-μέλη πλήρως να σέβονται την απαγόρευση αρνητικής μεταχείρισης με λόγο τις σεξουαλικές επιλογές είναι οι αρχές της μη αρνητικής μεταχείρισης ε, είναι ιερός ε, θα έλεγα θεμελιώδης νόμος, θεμελιώδης αρχή. Και όσον αφορά την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Το πρωτόκολλο για την εφαρμογή της χάρτας όσον αφορά την, ε, πρωτοβουλία της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τις δικαστικές αρχές και την ομολογία των χωρών αυτών αναφέρει ότι η χάρτα δεν επεκτείνει την ομολογία ή τις αρμοδιότητες ε, του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί δικαστηρίων της ε, Μεγάλου Βασιλείου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή της ε, Πολωνίας ώστε σε περίπτωση που βρίσκονται σε μη ευθυγραμμισμένες κάποιες αρχές με τις ελευθερίες, θεμελιώδεις ελευθερίες θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι ακριβώς ε, η οδός ώστε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ερμηνεύσει τα πρωτόκολλα αυτά αυτών των δύο κρατών μελών. Σα ευχαριστώ. Ashley Fox παρακαλώ. Πρόεδρε, Πολλέ χώρε ε, παγκόσμια έχουν σε σχέση με τα συντάγματα του ε, κάποιε τέτοιε αρχέ λιγότερε σε σχέση με την προστασία όμω των πολιτών του όσον αφορά αυτό θεωρείται ότι εδώ δεν πρόκειται για τη δομή των, ε, της προστασίας από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά για τον τρόπο εφαρμογής αυτών των, αρχών, των θεμελιωδών αρχών. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν εκλεγηγούν οι συντηρητικοί, θα αρνηθούν αυτές τις διατάξεις και θα την αντικαταστήσουν με μια άλλη διάταξη. Αυτό θα σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές για τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα εφαρμόζονται πλέον στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορείτε να εξηγήσετε λοιπόν σε σχέση με την προσυπογραφή το, της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς αυτό μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Η, το κόμμα μου θα ζητήσει και αλλαγή τη συνθήκης ώστε να, εγγυά, να εγγυόμαστε ότι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν θα έχει ε, οποιαδήποτε ανάμειξη με την ομολογία και τα νομικά θέματα στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς εσείς βλέπετε το θέμα, ευχαριστώ. Ήδη εν μέρει απάντησα το ερώτημα αυτό απαντώντα στην προηγούμενη τοποθέτηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλε χώρε έχουν ένα πρωτόκολλο που έχουν υπογράψει όσον αφορά την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έχουν το δικαίωμα αυτό. Το διαπραγματεύτηκαν, υπάρχει μια διακυβερνητική συνθήκη που αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Και αναφέρθηκε αυτό και έγινε αυτό, ενώ θα είχα προτιμήσει όλα τα κράτη-μέλη να είχαν υπογράψει και να είχαν αποδεχτεί τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διότι θεωρώ και πιστεύω ότι είναι θεμελιώδη πηξίδα αυτή η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Τώρα, σε σχέση με την πρόσβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτό θα ολοκληρώσει το πλαίσιο προστασία. Σέβομαι φυσικά το Ενωμένο Βασίλειο και το πλαίσιο το νομικό που υπάρχει για την ε, ασφάλιση των νομικών θεμάτων και των θεμάτων δημοκρατία πολυαίωνο μάλιστα. Και γι' αυτό θλίβομαι για το ότι δεν ανήκει ανήκει το Ηνωμένο Βασίλειο με τους υπόλοιπους εταίρους ε, στο να έχουν προσυπογράψει και να έχουν δεχθεί αυτό το γεγονός όπως οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Ε, Πέτρο, σας ευχαριστούμε. Η κυρία Φιγκερέδο, παρακαλώ. ήρθα Φιγκερέδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα δικαιώματα των γυναικών και το δικαίωμα να ζει κανεί μια ζωή με αξιοπρέπεια είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προωθούνται, να προάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λαμβάνοντα υπόψη τι ανισότητε που είναι κραυγαλέ και που συνεχίζουν να υπάρχουν και επιδεινώνονται κιόλα και οι ανισότητε οι μισθολογικέ μεταξύ ανδρών και γυναικών ακόμα τη φτώχεια. Η φτώχεια και η προσωρινή εργασία, η επισφαλής εργασία που πλήττει κυρίως ε, γυναίκες. Δεν φτάνει μόνο να διακηρύττουμε μια χάρτα δικαιωμάτων των γυναικών που είναι γενικόλογες αρχές ε, που δεν ε, σε σχέση με οποιαδήποτε συζήτηση με τις οργανώσεις γυναικών δεν έχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα ή σε σχέση και με την Ευρωβουλή. Γι' αυτό ερωτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη, είναι διαθέσιμη να δώσει προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών με συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα όμως ιδιαίτερα εξειδικευμένα στην εκπόνηση μιας νέας στρατηγικής για την ισότητα που το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζει μια έκθεση γι' αυτό ευχαριστώ και να πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Ευχαριστώ. Την προηγούμενη Παρασκευή με την κυρία Ρέντινγκ υπέβαλα μια πρόταση για τα δικαιώματα των γυναικών. Και έχουμε επίση την επιβεβαίωση από πλευρά τη Επιτροπή στη δέσμευσή μα αυτή και τη δέσμευσή μα και βούλησή μα να εργαστούμε προ αυτή την κατεύθυνση σε αυτό τον τομέα. Το Σεπτέμβριο αυτή η επιστολή που προαναγγείλαμε θα ακολουθηθεί από μια νέα στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό θα μα δώσει ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο θα είναι αρκετά ευρύ ώστε η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορέσει να πετύχει πρόοδο σε σχέση με τα δικαιώματα, ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως στα θέματα που αναφέρατε, από τη δουλειά και την απασχόληση μέχρι και άλλα θέματα που είναι σημαντικό να διασφαλιστεί αυτή η ισότητα για τις γυναίκες η, κάρτα, η, χάρτα αυτή θα πρέπει να εκφράζει και τις, ε, ε, τη διακήρυξη ε, μετά από 15 χρόνια της πλατφόρμας του Πεκίνου και να λαμβάνονται υπόψη οι διεκδικήσεις και από πλευράς των Ευρωβουλευτών που αφορούν τα θέματα των γυναικών. Και έτσι θα υπάρξει μία ακόμα συνεδρίαση, υπάρχουν τέτοιες συνεδριάσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι θα πετύχει αυτός ο στόχος. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Uh, το θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω σήμερα αφορά την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Το άρθρο 1.21 της Συνθήκης της Λισαβόνας ε, θα, προχωρήσει, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και ο λαός της Ελλάδας ε, είναι μεταξύ της Κύλας και της Χάραβης διότι τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ στη χώρα αυτή. Εσείς στείλατε τους ε, υπαλλήλους σας να διορθώσουν την κατάσταση. Θα γίνετε κυβερνήτης και της Ελλάδας. Αν ε, τα μέτρα τα οποία έχει περάσει η κυβέρνηση έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αν όχι, τι θα γίνει, θα φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Τι θα γίνει με άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι το θέμα μας σήμερα είναι η εφαρμογή της νέας συνθήκης και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό παρακαλώ να ε, παραμένετε στα πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος. Θέλετε να δώσετε μια απάντηση κύριε Πρόεδρε. Είμαι πάντα έτοιμος στις ερωτήσεις των μελών του Κοινοβουλίου, λέει ο Πρόεδρος Μπαρόσο. Το ερώτημά σας, αξιότιμο μέλος, προέρχεται από μια προϋπόθεση, θα έλεγα μια αρχική σκέψη που είναι λανθασμένη. Είναι σαν να λέτε ότι η Ελλάδα έχει προβλήματα επειδή είναι στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν πολλές χώρες εκτός της Ευρωζώνης που έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα και σε αρκετές περιπτώσεις πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Να σας θυμίσω τι συμβαίνει στην Ισλανδία, η οποία η Ισλανδία ζητάει να ενταχθεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζει κάποια στιγμή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον η Ισλανδία. Είναι εντελώς λάθος διανοητικά να πιστεύει κανείς ότι τα προβλήματα της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα επειδή δεν σεβάστηκε ακριβώς τους κανόνες της Ευρωζώνης αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες και ακριβώς πρέπει να πληρώσει το κόστος της δύσκολης προσαρμογής στην οποία πρέπει να προχωρήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέψτε μου μια ερώτηση για το πρόβλημα της αποθήκευσης δεδομένων, μια και το συνταγματικό δικαστήριο στη Γερμανία, την γενική αποθήκευση όλων αυτών των στοιχείων κατά την αρχή του μήνα την ακύρωσε. Εξακολουθεί να είναι επίμαχο το θέμα. Κατά πόσον ε, είναι εφικτή, ε, μπορεί να επιτρέπεται η αποθήκευση προσωπικών στοιχείων και αυτή είναι συμβατή και αν αυτό είναι συμβατό με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και εδώ θα πρέπει σε σχέση με συμφωνίες και σε σχέση και με την οδηγία για την αποθήκευση από της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνθήκη της Λισαβόνας ή στον κατάλογο της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνθήκης Λισαβόνας θα πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων για να αντιμετωπίσουμε την αποθήκευση δεδομένων. Έχει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα αυτό. Αν δηλαδή ο κατάλογος της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων ισχύει ή όχι. Ευχαριστώ. Η από προστασία των ε, θεμελιδών δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τι συνθήκε τη Λισαβόνα, μπορεί να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο τώρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για την προστασία τη ασφάλεια των πολιτών μα και για όλε τι διαδικασίε επεξεργασία ε, των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά εμπλεκόμαστε πλήρω στην αναθεώρηση αυτού του πλαισίου, μια και η διαδικασίε συναπόφαση επίση εφαρμόζεται για του στους τομείς του τρίτου πυλώνα. Επίσης πρέπει εξίσου να διασφαλίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών θα προστατεύονται όταν προσωπικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ σε σχέση με τη Συμφωνία για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ισχύει για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και το επεξεργαζόμαστε. Γίνονται διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η συμμετοχή των εμπλεκομένων και των πολιτών έχει υπόψη να υποβάλει μια πρόταση σύσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει επαρεξέταση των διαδικασιών και διεργασιών με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Κυρία Σάρα Λάτφορντ, Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας κατέστη δυσκολότερη λόγω των προβλημάτων σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λόγω και των πρακτικών της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ελπίζαμε με την κυβέρνηση Ομάπα, Ομπάμα συγγνώμη, τα πράγματα να αλλάξουν. Βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς συνεχίζονται τα στρατοδικεία ακόμα και αν κλείνει τον Γκουαντάναμο. Αυτές οι παραβιάσεις των διεθνών κανόνων καθιστούν τα προγράμματα ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε ακόμα πιο προβληματικά από ό,τι εμφανίζονται. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτές τις απαράδεκτες δικαστικές πρακτικές στις Ηνωμένε Πολιτείε. Σήμερα, ανεξάρτητα από αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν, δεν υπάρχει ο κίνδυνος στα πλαίσια της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη, εφόσον θυμάμαι καλά, που έθεσε το θέμα με τον πρόεδρο των, τέος πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου ακόμα και στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας όπως στην περίπτωση του Γκαντάναμο. Τότε εγώ και ο κύριος Σούσελ, πρωθυπουργός της Αυστρίας, είχαμε θέσει το θέμα. Και πάντα ζητούσαμε το θέμα αυτό να συζητιέται σε επίπεδο διαλόγου με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα εξακολουθήσει να συμβαίνει αυτό κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει όμως να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο είναι προαπαιτούμενο το κοινό αυτό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να βρούμε τον σωστό δρόμο, τον σωστό τρόπο να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν, την ανάγκη δηλαδή για το σεβασμό των ελευθεριών και την ανάγκη φυσικά για την ασφάλεια, γιατί αν δεν υπάρχει ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία. Η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα, ένα λεπτό. Ένα... από τα κύρια θέματα στη νέα συνθήκη Λισαβόνα είναι ο αυξημένο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πεδίο. Με αυτή την ενισχυμένη εξωτερική πολιτική, εμεί ω Ένωση πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο για την προαγωγή και υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτε χώρε. Ερωτήματά μου προ εμά είναι, τι κάνετε εσεί κύριε Μπαρόζο και κυρία Άστον, ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολιτική τη προαγωγή τη πολιτική υπέρ τη δημοκρατία. Δεύτερον, θα είσαστε υπέρ περισσότερων και μεγαλύτερων κονδυλίων για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον επόμενο προπολογισμό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα φαίνεται να παίρνουν επουσιώδη ρόλο να παίζουν ή και να έχουν τριτεύοντα ρόλο. Πρέπει όμω περισσότερο, περισσότερο χρόνο και κονδύλια να επενδύσουμε σε αυτά και να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα ταμείο για την δημοκρατία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Η διάταξη της συνθήκης ε, για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκόσμια έχει θεσπίσει τέτοιες αρχές η Ευρωπαϊκή Ένωση από την απαγόρευση της θανατικής ποινής ε, όπως και την υποστήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων από τις εξωτερικές ε, πολιτικές σχέσεις ή και διπλωματικά διαβήματα υπέρ αυτών των θεμάτων. Εγώ ίδιος έφυγα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνόδους κορυφής με εκπροσώπους από τρίτες χώρες. Πρόσφατα τώρα σε διάλογο που είχαμε υποβάλαμε και τονίσαμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύνοδο που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 40 τέτοια πλαίσια διαλόγων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκόσμια, καθώς επίσης και για τη διεξαγωγή των ε, ε, θεμάτων αυτών εξειδικευμένα. Για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 150 εκατομμύρια ευρώ διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη ΜΚΟ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσπαθούμε να εντάξουμε την ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε συμφωνία συνάπτουμε με τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σίμων Μπουσούτιλ, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία από τις θεμελιώδεις αρχές uh, που μας εμπνέει είναι η ελευθερία της uh, κίνησης και της ε, ελευθερίας κυκλοφορίας. Σε σχέση ακριβώς βλέπουμε με την ε, Λιβύη. Εκατοντάδες ε, πολίτες δεν μπορούν να εισέλθουν στην Λιβύη για να εργαστούν. Ερώτησή μου, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αναζητηθεί μια ε, λύση, μια δυνατότητα διεξόδου σε αυτό το πρόβλημα. Είναι αποδεκτό μια χώρα όπως η Ελβετία για παράδειγμα μονομερός να υιοθετεί μια απόφαση η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους πολίτες της ζώνης Σέγγεν και ιδιαίτερα για εκείνους τους εργαζόμενους που θα ήθελαν να απασχοληθούν, να εργαστούν ε, στην Λιβύη. Πρόεδρος, μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή η περίπτωση από πλευράς Επιτρόπου Μάνστρομ αναφέρθηκε ότι η ακύρωση δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας για τους πολίτες της ζώνης Σέγγεν δημιουργεί προβλήματα και υπάρχει θέμα το οποίο τίθεται στις σχέσεις μεταξύ Λιβύης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονα διπλωματικά διαβήματα βρίσκονται υπό εξέλιξη για να αναζητηθεί μια λύση. Για παράδειγμα, σε σχέση και με τους ε, Ελβετούς υπηκόους ε, που αντιμετώπισαν άμεσα προβλήματα. Και εδώ έχει υποστηρίξει η συνέχιση αυτών των διπλωματικών προσπαθειών και διαβημάτων. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάλογος ώστε να αναζητηθεί μια κατανόηση μεταξύ των συμβαλωμένων μερών και να αναζητηθεί μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο Λε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και τώρα εγώ θα ήθελα μεταξύ άλλων να πω ότι μέσα, μέσω της επικύρωσης της συνθήκης Λισαβόνας ο σεβασμός των θεμεριωδών δικαιωμάτων ενισχύθηκε. Όμως πέρυσι όταν Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την ομολογία του απέδειξε ότι τα δικαιώματα των συνδικάτων και των εργαζομένων πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο σε σχέση με την απόφαση Λαβάλ και Viking. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν τα έλαβε ακριβώς υπόψη όπως θα έπρεπε και το κατέστησε ανέφικτο και αδύνατο ώστε τα συνδικάτα να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και ίδιο μισθό μισθό για ίδια εργασία, άσχετα αν προέρχονται από το εξωτερικό ή είναι ε, εργάτες μιας ε, χώρας. Και από πλευράς ε, Επιτροπής ε, υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις που είχαν τότε γίνει σε εμά. Γι' αυτό η ερώτησή είναι προς εμάς κύριε Μπαρόζο. Πότε αναμένεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση ώστε αυτό το πρόβλημα να επιληθεί, το οποίο μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, δημιουργήθηκε. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να μας αναφέρει μια ημερομηνία σχετικά. Όταν δημοσιοποιήθηκαν αυτές οι αποφάσεις τοποθετηθήκαμε και εμεί σαφέστατα. Και εγώ και ο τότε Επίτροπος Σπίτλα που ήταν υπεύθυνο για την απασχόληση. Δηλαδή αποσαφηνίσαμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν μπορούν να αναθεωρήσουν θεμελιώδη δικαιώματα όπω το δικαίωμα ε, απεργίας, του συνδικαλίζεστε, άλλες ιδιομορφίες, εργασιακών σχέσεων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε κάποιες προτάσεις. Δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, δεν περίμενα αυτή την ερώτηση, ε, αλλά όπως σας είπα και κατά το παρελθόν, κατά την εκλογή αυτής της Επιτροπής, αυτό είναι ένα θέμα που, με το οποίο θα ασχοληθούμε άμεσα. Σας ευχαριστώ, κύριο Λιμπεράσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Ε, θεμελιώδεις αρχές, νέα συνθήκη, εξωτερική δράση. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, υπήρξαν κάποιες ε, ανεπαρκείς ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές. πώς η νέα συνθήκη θα βιώσει τον αριθμό σφαλμάτων κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού 33% ε, δημοσιονομικά σφάλματα έχουμε αυτή τη στιγμή. Πώς θα διορθωθεί αυτό. Όπως ξέρετε έχουμε προσπαθήσει χρόνια να μειώσουμε τα δημοσιονομικά σφάλματα στους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά από αυτά τα σφάλματα, όπως γνωρίζετε, οφείλονται στα κράτη-μέλη και στην εφαρμογή πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αισθάνομαι θετικά μετά τη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου που αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα δεν πρέπει να παραμένουμε αδρανείς. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για να μειώσουμε τα δημοσιονομικά σφάλματα που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή του προϋπολογισμού. David Κάσα, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, η συνθήκη αναφέρεται πώς διασφαλίζουμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν πρέπει να συμμορφώνονται με όσα ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έπραξε η Μάλτα και πολλές άλλες χώρες που γίνανε μέλη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στην Τουρκία. Όσον αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, πιστεύετε ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει ακόμη πολλά πράγματα κύριε Πρόεδρε και τι θα κάνει η Κομισιόν ώστε να εξασφαλίσει ότι προτού σταθεροποιηθεί η οικονομία της και προτού συμμορφωθεί η Τουρκία γενικότερα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα θα προστατευτούν ενώ είναι ανύπαρκτα στην Τουρκία σήμερα. Δεν θα έλεγα ανύπαρκτα, λέει ο κ. Μπαρόζο, να είμαστε ειλικρινεί. Η πρόοδο έχει εξελιχθεί όσον αφορά το κράτο δικαίου. Δεν πιστεύουμε ότι έχει φτάσει στο επίπεδο σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων στο επίπεδο του ευρωπαϊκού. δεν έχει φτάσει ακόμη. Θα χρειαστούν χρόνια. κάθε χρόνο, επειδή είναι υποψήφια χώρα η Τουρκία ή η Κομισιόν, ε, αξιολογεί πολύ αντικειμενικά τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το ε, κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έχουν υπάρξει πρόοδοι, να είμαστε δίκαιοι. Βεβαίω υπάρχουν και άλλα θέματα για τα οποία οι τουρκικές αρχές πρέπει να εργαστούν περαιτέρω ο διάλογος και αυτές οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας ουσιαστικά διασφαλίζουν πρόοδο όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής μεταρρύθμισης στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μια ουσιαστική συνάντηση. Η επόμενη θα γίνει σε ένα μήνα την επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου. Ευχαριστώ πολύ. It is end of our discussion. Τελειώνει η πρώτη μας αυτή συζήτηση. Το επόμενο θέμα είναι η διεθνής πολιτική για τις κλιματολογικές αλλαγές. E- Κυρία Πρόεδρε, ακούστηκα προηγουμένως σε αυτή την αίθουσα κάποια φοβερά πράγματα εις βάρος του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι το Προεδρείο του Σώματος δεν θα πρέπει να επιτρέψει να συζητιώνται θέματα εθνικής πολιτικής σε αυτή την Ολομέλεια. Όταν συχνά πρόκειται για θέσματα συνταγματικά και θετικά πολύ μεγάλη σημασίας, και θυμίζω σε όλους τους συναδέλφους ότι η Ιταλική Δημοκρατία δεν είναι προσπόληση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Τζόρτζο Ναπολιτάνο, είναι ο θεματοφύλακας του Ιταλικού Συντάγματος. Εξ ονόματος λοιπόν της Ιταλικής Συνιστώσας, του Σοσιαλιστικής Ομάδας, θα ήθελα να καλέσω την Προεδρία του Κοινοβουλίου να είναι πιο προσεκτική σε σχέση με τα θέματα τα οποία επιλέγονται να συζητηθούν και στις ομιλίες οι οποίες γίνονται. Λυπάμαι που ο πρόεδρος κ. Μπούζεκ δεν πήρε το λόγο έτσι ώστε να διακόψει μία ξεκάθαρη επίθεση εις βάρος του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας ο οποίος ε, πριν μια εβδομάδα επισκέφθηκε επίσημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ähm, Ευχαριστώ θερμά και αυτά που αναφέρατε φυσικά στα πρακτικά θα καταχωρηθούν πλήρως και θα προσπαθήσω για το σημείο της ημερήσιας διάταξης για το οποίο είμαι αρμόδια να ανταποκριθώ στα αιτήματά σας. Το ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Αξιότιμοι συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη